Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το υπαριθμόν 12. Οι συστάσεις των συντονιστών έχουν δυναμηθεί ηλεκτρονικά. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούν, μπορεί να θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν και μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 13 της ημερησίας διάταξής μας, που είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του σωριστικού κόστους στη χημική βιομηχανία, στο πλαίσιο του Ρεφίτ. Και θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Πετινέλη, να πάρει το λόγο και να μας εξηγήσει τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους αυροβουλευτές που με καλέσατε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω το πλαίσιο και κάποια πρώτα ευρήματα της μελέτης μας σχετικά με ε, το σωρευτικό κόστος στη χημική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελική εκδοχή της μελέτης ε, θα δημοσιευτεί στην ε, ιστοσελίδα μας ε, μετά από την επικύρωσή της. Πρόκειται για μελέτη που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε παροχό υπηρεσιών χρησιμοποιώντας έγκυρη μεθοδολογία. Η μελέτη αυτή αποτελεί σημαντικά στοιχεία για τη δουλειά μας. Δεν είναι όμως μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα χημικά είναι απαραίτητα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον. Αδιαμφισβήτητα είναι απαραίτητη η νομοθεσία στον τομέα των χημικών και είναι προφανή τα ωφέλη της νομοθεσίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η νομοθεσία και ε, την ε, οικονομική βιωσιμότητα ε, της χημικής βιομηχανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό αναθέσαμε σε σχετικό φορέα να εξετάσει το σωρευτικό κόστος στη χημική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση του σωρευτικού κόστους επικεντρώνεται στο κόστος και όχι σε άλλες συνέπειες της νομοθεσίας. Έτσι, η μελέτη αυτή δεν θα πρέπει να εξεταστεί απομονωμένα, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει οικοδομικό λίθο για την καλύτερη κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματοποιούνται άλλες μελέτες σχετικά με το πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα ωφέλη της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ε, και κάποια δεδομένη στιγμή θα εξεταστούν μαζί όλα τα ευρήματα. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν ε, την αξιολόγηση και θα σας εξηγήσω και την σχέση ανάμεσα στη μελέτη αυτή και σε άλλες σχετικές μελέτες. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ καλά την διαφάνεια. Υπάρχουν διάφοροι τομείς στην χημική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, άλλοι είναι μεγάλοι, άλλοι μικρότεροι και συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο ε, στην οικονομία και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχει μεγάλος, ε, μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων ε, που αφορά την χημική βιομηχανία. Και γι' αυτό έχουμε χωρίσει εδώ την νομοθεσία στους διάφορους τομείς που βλέπετε στις διάφορες στήλες. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στους τομείς που είναι πιο αντιπροσωπευτικοί και για τους οποίους ήταν δυνατόν να συλλέξουμε επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία είναι οι τομεί που βλέπετε με γαλάζιο, ενώ δεν έχουμε εξετάσει τους ε, λευκούς ε, τομείς εδώ πέρα. Ε, θα έχετε στη διάθεσή σας μετά την παρουσίασή μου τις διαφάνειες αυτές. Και περνώ στην επόμενη διαφάνεια να σας παρουσιάσω τα πρώτα ευρήματα της μελέτης μας εξέλιξη του κόστους στο διάστημα 2004-2014. Η εξέταση του κόστους δείχνει ότι αυξάνεται το ρυθμιστικό κόστος. Ε, είδαμε σημαντικές αυξήσεις ε, από το 2007 στο 2008 λόγω ε, της θέσης σε ισχύ του REACH και του CLP και ε, επίσης ε, βλέπουμε αργότερα παρόμοια ε, αύξηση. Είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ο υπολογισμός, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδέσουμε την αύξηση του κόστους με συγκεκριμένα νομοθετήματα. Κάποια μέρη του κόστους εμφανίζονται αμέσως, ενώ άλλα εμφανίζονται σε βάθος χρόνου. Τρεις ε, βασικές αιτίες υπάρχουν ε, ε, για το κόστος. Το 1 τρίτο συνδέεται με τις εκπομπές το άλλο τρίτο συνδέεται με την ε, νομοθεσία περί χημικών και το τρίτο τρίτο ε, από την νομοθεσία για την ασφάλεια των εργαζομένων. Και δεν είναι μόνο το REACH ε, η σχετική νομοθεσία που έχει επιπτώσεις στο κόστος. Δεν ε, μπορούν ε, όλα τα ερωτήματα να απαντηθούν ε, στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης του σωρευτικού κόστους. Θα πρέπει κάποιες από τις δαπάνε να εξεταστούν ξεχωριστά. Άλλο αποτέλεσμα της μελέτης που είναι ενδιαφέρον έχει να κάνει με την προστιθέμενη αξία σε διάφορους τομείς. Για τα ζύζαν και άλλα χημικά βλέπουμε ότι το νομοθετικό κόστος ε, ανέρχεται στο 30% ενώ σε άλλους τομεί είναι πολύ πιο χαμηλό όπως για παράδειγμα στα πλαστικά. Ε, το κόστος αυτό ε, επηρεάζει την οικονομική βιωσιμότητα των εταιριών και γι' αυτό και τη δυνατότητά τους να επενδύσουν στο μέλλον. Γι' αυτό και μάλιστα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι ανταγωνιστές τους δεν πληρώνουν ανάλογο κόστος. Ε, δεν μπορούν όμως ε, από τη μελέτη αυτή να ε, εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με, το αν, με την καταλληλότητα της νομοθεσίας μας. Αυτό θα φανεί από το fitness check, τον έλεγχο καταλληλότητας. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω καλύτερα ε, το, το διαφορετικό στόχο ε, ανάμεσα ε, στις δύο αυτές αξιολογήσεις. Την αξιολόγηση του σωρευτικού κόστους, το CCA και το fitness check, τον έλεγχο καταλληλότητας. Εξετάζουμε εμείς το σωρευτικό κόστος για την βιομηχανία χημικών, ενώ ο έλεγχος καταλληλότητας εξετάζει την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα ε, και σκοπιμότητα ε, της νομοθεσίας. Ε, άλλο δηλαδή να εξετάζουμε την ε, νομοθεσία και άλλο τώρα εξετάζουμε το σχετικό βιομηχανικό τομέα. Η μελέτη μας βασίστηκε σε μεθοδολογία που στόχο έχει να αναλύσει τις συνέπειες της νομοθεσίας στην βιομηχανία χημικών. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στον έλεγχο καταλληλότητας για την νομοθεσία πέρα από το ΡΙΤΣ. Το ξεχωριστά για να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική από την ανάλυση αυτή, θα πρέπει να εξετάσουμε ποιο κόστος είναι σημαντικό όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ε, νομοθεσίας περιχημικών. Θα πρέπει να αποφύγουμε άμεση σύγκριση ανάμεσα σνικά ωφέλη της νέας νομοθεσίας ε, με το ε, κόστος των επιχειρήσεων, διότι μπορεί το κόστος αυτό να είναι εις βάρος της κοινωνίας, ε, για παράδειγμα όταν οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας. Ωστόσο θα πρέπει να εξεταστούν ε, οι συνέπειες κατά περίπτωση. Ε, έτσι λοιπόν έχουμε μια δεύτερη φάση της ε, μελέτης μας ε, όπου εξετάζουμε τις διαφορές ανάμεσα στο κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα μέρη του κόσμου για να δούμε εάν υπάρχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας παρακαλούσα να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος. θα ε, συμπληρώσουμε τη μελέτη μας με μια δεύτερη φάση όπου εξετάζουμε τη ε, διαφορά ανάμεσα στα σχετικά κόστη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε άλλες περιοχές του κόσμου, του κόσμου για να δούμε εάν οδηγούν σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξετάσουμε τη σκοπιμότητα της νομοθεσίας μας. Ήδη τα αποτελέσματα της μελέτης μας ε, μπορούν να εξεταστούν ε, για να ε, δούμε μήπως μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στην νομοθεσία μας. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος αυτό χωρίς να μειώσουμε το επίπεδο προστασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας περί χημικών και στο πλαίσιο της οικονομικής βιωσιμότητας οποιασδήποτε εταιρείας. Συμπέρασμα. Ο βασικός μας ε, στόχος ε, είναι να διαπιστώσουμε ε, πού βρίσκονται τα όρια της οικονομικής βιωσιμότητας σε σχέση με την νομοθεσία περί χημικών μας. Τώρα λοιπόν έχουμε στοιχεία στη διάθεσή μας και είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι εργασίες και να εξετάσουμε το ρυθμιστικό κόστος στο ευρύτερο πλαίσιο. Να εξετάσουμε δηλαδή την προστιθέμενη αξία το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να θεωρηθεί σχετικά χαμηλό, μπορεί όμως να εξαντλεί ε, τα οικονομικά ε, αποθέματα, τα οποία θα, πρέπει, θα, θα ήταν προτιμότερο να επενδύσουμε στην έρευνα και καινοτομία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. και τώρα δεν ξέρω αν ε, κάποια από τα μέλη θέλουν να κάνουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είπε ότι η έρευνα CCA είναι το κομμάτι ενός παζλ της νομοθεσίας. Αυτό όμως το οποίο δεν καταλαβαίνω εγώ είναι ένα πράγμα το αν σε αυτήν την, θα λέγαμε, εμπορική έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στην επιρροή της νομοθεσίας στη χημική ε, βιομηχανία, αν θελήσατε να εντοπίσετε το πώς η χημική βιομηχανία Ε, έχει κόστος για, την, για τον εθνικό προϋπολογισμό και με την απουσία νομοθεσίας τότε δεν θα έχει κόστος στον προϋπολογισμό διότι ε, αυτό δεν θα συνέβαινε πιστεύω. Ε, αν δεν νομοθετούμε λοιπόν τότε θα έχουμε υψηλότερα κόστη για την υγεία για παράδειγμα. Οπότε αναρωτιέμαι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει το αν η χημική βιομηχανία δεν προκαλεί επιπλέον κόστη στους ε, δημοσίους προϋπολογισμούς και ένα ακόμα θέμα το οποίο με εκπλήσει υπόθηκε ότι είναι μια μη δεσμευτική έρευνα όμως κάτι τέτοιο είναι πολύ γενικό λόγο και με κάνει να αναρωτιέμαι πόσο έχει κοστίσει εφόσον είναι μη δεσμευτική. Ο κύριος Όσλινγκ. Ναι, θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο, διότι το ερώτημα αφορά ε, την ανταγωνιστικότητα για την ε, χημική βιομηχανία. Αυτό είναι, όμως, ε, αυτό είναι ένα θέμα. Όμως, από την άλλη, είναι λογικό να δίνουμε την εντολή για μια τέτοια έρευνα η οποία δεν εξετάζει αυτά τα οποία είπε ο προηγούμενος συνάδελφος. Όπως είναι, για παράδειγμα, τις την ε, ε, αποτροπή ε, υγειονομικών κοστών λόγω μιας καλής νομοθεσίας. Αυτό δεν υπάρχει στην έρευνά σας. Ναι, υπάρχει το κόστος σχετικά με την νομοθέτηση, όμως όσον αφορά το γενικότερο θέμα λέμε ότι θα πρέπει να μειωθεί η νομοθεσία διότι αυτό περιορίζει τη βιομηχανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται διότι η χημική βιομηχανία ε, ε, ε, δεν τα πηγαίνει καλά λόγω της υπερβολικής νομοθεσίας. Συγγνώμη αν να το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό. Και γι' αυτό το λόγο το ερώτημα μου είναι αν θα επακολουθήσει και άλλη μια έρευνα η οποία να αναφέρει και τα θετικά της νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Διότι έχουμε νομοθεσία η οποία όπως κατάλαβα προκαλεί μεγάλη κόστη, όμως σίγουρα θα έχει και ωφέλη και ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας όταν δηλαδή συνυπολογίζουμε μαζί μας το κόστος για το περιβάλλον για παράδειγμα. Αυτό το οποίο θα με ενδιαφέρει επιπλέον είναι τι βάση δεδομένων χρησιμοποιήσατε, είχατε στατιστικά δεδομένα, όμως ε, δεν αναφερθήκατε συγκεκριμένα που αναφέρετε, οπότε λυπάμαι, αλλά θεωρώ ότι η Επιτροπή έχει μια ξεκάθαρη στάση. Ε, θεωρώ τη διαδικασία αυτή ε, πολύ γενική και δεν νομίζω λοιπόν ότι ταιριάζει επαρκώς και δεν νομίζω ότι βοηθάει επαρκώς την επίλυση του προβλήματος. άλλες ερωτήσει, όχι. Οπότε μπορούμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να δώσει απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τη μελέτη αυτή καθεαυτή, όπως είπα στην αρχή της παρέμβασής μου, η μελέτη αυτή αποτελεί στοιχείο μιας γενικότερης αξιολόγησης που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε τον πέμπτο έλεγχο REFIT, την πέμπτη αξιολόγηση όσον αφορά την βελτίωση της νομοθεσίας, όπου θα προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε όλα τα ωφέλη, όλη τη μείωση κόστου σε εθνικό επίπεδο μέσω της νομοθεσίας REACH και άλλης νομοθεσίας που έχει να κάνει με τη χημική βιομηχανία. Περαιτέρω αξιολόγηση επίσης νομοθεσίας REACH θα γίνει γιατί αυτό προβλέπεται και στον ίδιο τον κανονισμό. Μόνο όταν θα έχουμε λοιπόν μια σφαιρική εικόνα θα είμαστε θέση να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Όπω είπα άλλωστε και στην αρχή τη παρεμβασή μου, βρισκόμαστε μόνο στην αρχή τη όλη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα την μελέτη αυτή καθεαυτή, όπω και για κάθε μελέτη που γίνεται από φορείς οι οποίοι δικαιεύονται σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους τομείς όπως η χημική βιομηχανία, η ε, έρευνα αυτή έχει ως στόχο όχι τόσο πολύ να καταλήξει συμπεράσματα, αλλά περισσότερο να ενημερώσει, να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτό ακριβώς εμείς ζητήσαμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον εξωτερικό φορέα που ανέλαβε αυτή την έρευνα. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποσοτικά ποιο είναι το σωρευτικό κόστος στη χημική βιομηχανία. Δεν εναπόκειται όμως στον ε, φορέα έρευνα ε, να καταλήξει συμπεράσματα. Μα παρέχει απλώ κάποιε πληροφορίε και εμεί συνέχεια ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογούμε αυτέ τι πληροφορίε και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε κάποιε συστάσει προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τώρα το κόστο τη έρευνα, νομίζω ότι ήταν 350.000 ευρώ. Και αν δεν κάνω λάθος κατά αυτόν τον τρόπο, απάντησα και στο σύνολο των ερωτήσεών σας. Για άλλη μια φορά όμως θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για ένα μόνο συστατικό στοιχείο έρευνα αυτή που θα συμβάλλει τελικά στην αξιολόγηση REFIT στα πλαίσια της οποίας θα μας σε να δούμε αν όντω η υφιστάμενη νομοθεσία είναι η καλύτερη δυνατή. Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη από την ύπαρξη μιας νομοθεσίας όσον αφορά το χημικό τομέα. Επ' αυτού δεν τίθεται καμία αμφιβολία. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε. Ο κύριος Χόισλινγκ θέλει το λόγο, παρακαλώ. Äh, Δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου σχετικά με τη στατιστική βάση της μελέτης. Από πού προέρχονται τα δεδομένα. Είναι στοιχεία της ίδιας της χημικής βιομηχανίας. Πρωτού απαντήσετε ε, να ακούσουμε και την παρέμβαση του κυρίου Πότς. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Μία συμπληρωματική ερώτηση έχω. Πάντα θεωρούσα ότι η μελέτη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το JRC. Γιατί ανατέθηκε εξωτερικά η μελέτη αυτή τη στιγμή που έχουμε το JRC, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο πάντα είναι ε, ικανή να κάνει μια τέτοια μελέτη και νομίζω πήρατε 350.000 ευρώ για μια μελέτη την οποία θα μπορούσε να έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να, απαντήσω από την ε, να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. να διευκρινίσω ότι όταν αναθέτουμε μια μελέτη ε, στο JRC, στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, ε, πάλι πρέπει να μεταφέρουμε χρήματα, δεν γίνεται δωρεάν. Δηλαδή τα χρήματα μεταφέρονται είτε στο JSC είτε σε κάποιον ε, εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Η μελέτη ανατέθηκε με την κανονική διαδικασία ανάθεση. έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, δεν έχω λοιπόν όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ανατέθηκε με τις ε, διαδικασίες περί δημοσίων διαγωνισμών. Ε, αλλά επαναλαμβάνω όμως ότι και το JRC πληρώνεται, οπότε οικονομικά δεν υπήρχε καμία διαφορά. Όσον αφορά την μεθοδολογία, δεν υπάρχουν ε, στατιστικές στον τομέα αυτών. Έτσι λοιπόν, ο, φορέας που έκανε τη μελέτη ζήτησε τα στοιχεία από τις σχετικές βιομηχανίες. Οι επιχειρήσεις λοιπόν έχουν παράσχει τα στοιχεία. Έχουν χρησιμοποιηθεί εσωτερικά λογιστικά στοιχεία από τις εταιρείε. Είναι τα καλύτερα τα στοιχεία που μπορούσαμε να λάβουμε. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα καλύτερα στοιχεία. Δεν ε, διατίθενται κανονικά τα στατιστικά αυτά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι είναι ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί. Και τώρα μπορούμε να κλείσουμε εδώ με αυτό το σημείο της ε, ημερησίας διάταξης και να, και να περάσουμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε την Κομισιόν που βρισκόταν <coughs> εδώ. Μπορούμε λοιπόν να πάμε στο επόμενο που αφορά την ε, παρουσίαση, την παρουσίαση για την εγκληματικότητα κατά των Γριονιδών. Έχουμε εδώ την ε, κυρία ε, Γκέρ και τον κύριο Σίνα από το Ecologic Institute ε, για να παρουσιάσουν την έρευνα. Έχει 10 λεπτά ο καθένας. Έχετε το λόγο και μπορείτε να ξεκινήσετε με την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτήν την εισαγωγή ε, να παρουσιάσω τη συγκεκριμένη έρευνα στο κοινό σας. Προερχόμαστε και οι δύο από το Ecologic ε, ε, Institute, το οποίο βρίσκεται στο Βερολίνο. Όπως βλέπετε και στην παρουσίαση, αποτελούμαστε από αρκετά Ινστιτούτα. Στόχος ε, της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να παράσχει μια ε, γενικότερη εικόνα σχετικά με την εγκληματικότητα κατά των αγρίων ειδών στην Ευρώπη και τον ρόλο όσον αφορά την ε, εφαρμογή του συγκεκριμένου θέματος αλλά και ε, την προστιθέμενη αξία της προστασίας άγριων ειδών που όπως γνωρίζετε υιοθετήθηκε από την, ε, από την Κομισιόν στις 26 Φεβρουαρίου. Τώρα κάποια πράγματα όσον αφορά την μέθοδο που χρησιμοποιούσαμε στη συγκεκριμένη έρευνα. Φυσικά και εξετάσαμε την ακαδημαϊκή και επίσημη λογοτεχνία. Κάναμε μια ε, ιντερνετική έρευνα σε 25 κράτη-μέλη, όμως δυστυχώς λάβαμε ελάχιστες απαντήσεις. Επιπρόσθετα είχαμε μια σύνθεση δεδομένων από τη βάση δεδομένων EUTWIX, η οποία κεντροποιεί τα δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια κάναμε μία εις βάθος ε, ανάλυση χωρών και συγκεκριμένα έρευνε, ε, συνεντεύξεις ε, με πέντε χώρες συγκεκριμένοι, συγκεκριμένα Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συγκεκριμένες αναφορές για τις χώρες δημοσιεύθηκαν χωριστά από την συγκεκριμένη έρευνα και στη συνέχεια είχαμε ορισμένες προτάσεις οι οποίες εξελίχθηκαν κυρίως με βάση δικά μας ευρήματα αλλά και βασιζόμενοι και σε άλλα ευρήματα όπως είναι για παράδειγμα αυτά από το πρόγραμμα e-Face το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και ορισμένα από τα μέλη της έρευνας αυτής ε, συμμετείχαν επίσης στη συγκεκριμένη έρευνα. Τώρα, πολύ ε, σύντομα, θα προσπαθήσω να σας δείξω μια γενικότερη εικόνα ε, των συμπερασμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο προορισμός, αλλά και μια περιοχή τράνσιτ ε, για άγρια ζώα. Ως τράνσιτ έχει προβλήματα όσον αφορά τα θηλαστικά, ενώ ως προορισμός αφορά τα ερπετά, το χαβιάρι, ε, παπαγό, παπαγάλους και εναλλακτικά ιατρικά προϊόντα. Η, ε, ε, επικεντρωνόμαστε σε Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά ε, τις συγκεκριμένες ε, αποστολές ε, και, όλο και περισσότερη σημασία έχουν τα ταχυδρομικά κέντρα και φυσικά το ίντερνετ όσον αφορά την αποστολή των συγκεκριμένων ειδών. Στη συγκεκριμένη έρευνα ταυτοποιήσαμε τέσσερις βασικές διαδρομές εμπορίου. Αρχικά τα μεγάλα θηλαστικά όπως ε, ρινόκεροι, ελέφαντες, μέσω της Αφρικής και της Νότιας δικτύου Αμερική ε, φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι, μέσω εμπορικών κέντρων. Ε, στη συνέχεια έχουμε ε, παράκτια, παράνομη διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχουμε και απειλούμενα είδη πτηνών από την νοτιοανατολική Ευρώπη προς την νότια Ευρώπη, ενώ έχουμε και ρωσικά άγρια τα οποία εισάγονται μέσω των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών ενώ επίσης έχουμε και εισαγωγές εναλλακτικών ιατρικών προϊόντων τα οποία προέρχονται από τα θηλαστικά τα οποία ε, εισάγονται από την Ασία και στη συνέχεια επιστρέφονται ως ε, ιατρικά προϊόντα με την Ευρώπη ως ε, προορισμό. Όσον αφορά τα ρωσικά είδη, εκεί είναι πιο πολύπλοκο το θέμα, διότι δεν έχουμε ακριβή γνώση σχετικά με την ε, χώρα στόχο και μπορείτε να δείτε τις διαδρομές τα κόκκινα βέλη αφορούν την πρώτη κατηγορία ε, που αφορά δέρματα ζώων και ελεφαντόδοντο. Το πράσινο αφορά ε, το παράκτιο εμπόριο. Το πράσινο μετά αφορά τα πτηνά και το γαλαζοπό αφορά ε, τα ρωσικά άγρια είδη. Τώρα όσον αφορά την νομοθεσία και την εφαρμογή αυτής, ε, το νομοθετικό πλαίσιο κρίνεται γενικότερα επαρκές και η βασική ε, ανησυχία είναι η ελλειπής, η άνηση εφαρμογή του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ συχνά υπάρχει ένα περιορισμένο ή χαμηλό επίπεδο κυρώσεων, έλλειψη τεχνικών γνώσεων, αντίληψη τη κατάστασης, ειδίκευση ε, για την ε, από την πλευρά της αστυνομίας, ε, των εισαγγελέων ε, και επιπρόσθετα δίνεται περιορισμένη προτεραιότητα όσον αφορά την εγκληματικότητα κατά τον άγριο ειδών. Επίσης έχουμε ελάχιστη πληροφόρηση από την πλευρά των κρατών πελών όσον αφορά τι κυρώσει, ε, η, οποία η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τα κράτη-μέλη και επίσης έχουμε ελάχιστη πληροφόρηση όσον αφορά το επίπεδο και την ποιότητα της συνεργασία μεταξύ των αρχών τόσο ε, στο εσωτερικό αλλά και σε διεθνέ επίπεδο όσον αφορά τώρα το οργανωμένο έγκλημα και το ε, εξέπλυμα μαύρου χρήματος. και εκεί η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τα κράτη-μέλη. Σε πάρα πολλά κράτη-μέλη λοιπόν δεν λάβαμε καθόλου αποδείξεις ε, σχετικά με την κατάσταση, όμως και πάλι έχουμε ελάχιστα εμπειρικά δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, η προστιθέμενη αξία ε, για ένα σχέδιο δράσης πάνω στην εγκληματικότητα ε, κατά των άγριων ειδών είναι ε, στη διαδικασία των ε, συζητήσεων. Τώρα θα ήθελα να σας δώσω μια γενικότερη εικόνα σχετικά με τις προτάσεις που κάνουμε με βάση ε, τα ζητήματα. Αρχικά την, το ζήτημα προτεραιοτήτων. Αποτελεί προϋπόθεση για την επαρκή κατανομή πόρων αυτό είναι σημαντικό τόσο σε πολιτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το πολιτικό επίπεδο είναι σημαντικό όχι μονάχα να μιλάμε για ελέφαντες και ειρηνό και ρούσα, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και τα άλλα φυτά και ζώα τα οποία συμπεριλαμβάνονται, όπως είναι για παράδειγμα τα ερπετά. Και ένα άλλο ζήτημα προτεραιότητας είναι να κάνουμε την καλύτερη χρήση των περιορισμένων μέσων, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας, ε, το ελέγχους. Ένα άλλο θέμα είναι η μείωση της ζήτηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνουμε να αναγνωρίσουμε στρατηγικέ στρατηγικές ε, για την ε, μείωση ε, της ζήτησης και από την άλλη πλευρά να υποστηρίξουμε τις ε, δραστηριότητες για την μείωση της ζήτησης σε χώρες καταναλωτές. Ε, η δίκευση είναι ένα άλλο θέμα. Προτείνουμε να υπάρξει εκπαίδευση σε εξειδικευμένο προσωπικό Η συνεργασία τώρα είναι επίσης ένα άλλο θέμα θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενασχόληση από την πλευρά της Eurojust και της Europol. Θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των διασυνεργειακών δραστηριοτήτων και να υπάρξει χρηματοδότηση σημαντικών ε, παραγόντων όπως είναι για παράδειγμα τα δίκτυα στην όπνευση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η καταγραφή δεδομένων και πρόσβαση σε αυτά το οποίο είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε στοχευμένους ελέγχους και επιπρόσθετα συστήνουμε να να, να ε, προτείνουμε ή μάλλον και να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν το ζήτημα της ανταλλογής δεδομένων τώρα όσον αφορά τις κυρώσεις ε, οι ε, κυρώσεις θα πρέπει να αντεκατοπτρίζουν τη σοβαρότητα του εγκλήματος προτείνουμε στα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ε, μια ε, προσέγγιση εργαλειοθήκης, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν διάφορα μέσα όπως είναι ε, για παράδειγμα το ποινικό δίκαιο αλλά και διοικητικέ κυρώσεις, ενώ άλλο ένα θέμα είναι η εναρμόνιση των κυρώσεων, το οποίο είναι ένα δύσκολο θέμα, το οποίο απαιτεί αρκετή συζήτηση. Αν όμως κανείς σκεφτεί ε, την εναρμόνιση, τότε θα πρέπει να το σκεφτεί στο πλαίσιο της οδηγίας ε, για το περιβαλλοντικό έγκλημα. Θα κλείσω την παρουσίασή μου τώρα με κάποια σχόλια με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε κάποιες προτάσεις στην έρευνά μας. Αρκετά σημεία ανταποκρίνονται με την μορφή ε, του σχεδίου δράσης το οποίο υιοθετήθηκε το Φεβάρι από την πλευρά της ε, Κομισιόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην, ε, στην, όχι μονάχα στην εφαρμογή αλλά και στην πρόληψη θα πρέπει να υπάρξει μια εισήγηση προς την πλευρά του Συμβουλίου και καλούμε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο θέμα και απαιτείται φυσικά ε, πολιτική προτεραιότητα. Δεν έχουμε, ε, να μην υπάρχει εναρμόνιση ε, των κυρώσεων μονάχα για εγκλήματα για άγρια είδη. Όσον αφορά τώρα τα μεμονωμένα μέτρη, υπάρχει μεγάλη σύγκληση μεταξύ των προτάσεών μας και το σχεδίο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να σημειώσω κάτι τελευταίο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ε, του σχεδίου δράσης, το οποίο ε, βασίζεται σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική δέσμευση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Ζαβόρ πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, μελέτη αυτή, για την παρουσίαση του πορίσματος της μελέτησης Ανήκω στην διακομματική ομάδα για τα άγρια είδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε να έχουμε τελικά ένα σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της εγκληματικότητα εις βάρος των άγρων ειδών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι τεράστιο επίτευγμα το ότι επιτέλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει ένα σχέδιο δράσης σχετικό. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντική πρόοδο. Μολονότι βέβαια Πιστεύω ότι το σχέδιο δράσης δεν είναι όσο φιλόδοξο θα μπορούσε να ήταν. Συμφωνώ με τα περισσότερα από τα πορίσματα της μελέτης σας και αν κατάλαβα καλά, εσείς αξιολογείτε την κατάσταση κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, λέτε ότι το εφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι καλό, και ότι α, ε, ταιριάζει τελικά στην υφιστάμενη κατάσταση και ότι αρκεί για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας κατά των άγρων ειδών. Συμφωνώ ότι στα πλαίσια του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της δράσης μας κατά της εγκληματικότητας εις βάρος των άγρων ειδών και αυτό μπορεί να γίνει με τα κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης, εξειδίκευσης, με καλύτερη χρηματοδότηση διαφόρων δράσεων και του ίδιου του προσωπικού, για προγράμματα κατάρτισης δηλαδή. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα χρειαστούν επιπλέον νομοθετικές πράξεις προκειμένου να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος των άγρων ειδών. Επίσης, στη μελέτη σας αναφερόμενοι στο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέτε ξεκάθαρα ότι η έλλειψη νομοθετικής εναρμόνισης και ότι δεν υπάρχουν αποτελεσματικές κυρώσεις σε επίπεδο κρατών μελών αποτελεί τεράστιο εμπόδιο στο να είναι τελικά πραγματικά αποτελεσματική η μάχη αυτή κατά της εγκληματικότητας εις φάρος των άγρων ειδών. Χρειάζεται λοιπόν μια εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό λειτουργικό σύστημα κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να μπορεί στην πράξη να μειώνει τα φαινόμενα εγκληματικότητα και να τιμωρεί τους υπετίους εγκληματικότητα κατά των άγρων ειδών. Επίσης, να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι ε, η εγκληματικότητα κατά των άγρων ειδών ή ε, το λαθρεμπόριο τέτοιων ειδών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο μεμονωμένο. Πολύ συχνά μιλάμε για συστηματική προσέγγιση, αλλά μην ξεχνάμε ότι η εγκληματικότητα αυτή κατά των άγρων ειδών συνδέεται άμεσα με άλλες ομάδες σοβαρού εγκλήματος, συνδέεται πολλές φορές με ομάδες που ειδικεύονται στο λαθρεμπόριο, στο λαθρεμπόριο όπλων, στην εμπορία ανθρώπων και το καθεξής. Συνεπώς θα πρέπει να αρμονίσουμε όχι μόνο τις δράσεις και την νομοθεσία των κρατών μελών ως προς την εγκληματικότητα κατά των άγρων ειδών, αλλά πρέπει εν γέννη να αρμονίσουμε τη δράση μας κατά άλλων μορφών εγκληματικότητας και άλλων μορφών ε, οργανωμένου εγκλήματος και σε άλλους δηλαδή τομείς. Ακριβώς επειδή, όπως σας είπα, όλες αυτές οι μορφές εγκληματικότητας συνδέονται η μία με την άλλη και πολλές φορές είναι ακριβώς οι ίδιες οι εγκληματικές ομάδες οι οποίες μπορεί να υποφελούνται από διακίνηση ναρκωτικών, για παράδειγμα, μπορεί παράλληλα να έχουν προσόδους και από εγκλήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη διακίνηση άγρων ειδών. Και κάτι ακόμα, ένα ακόμα ζήτημα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι το ζήτημα της διαφθοράς. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καταρτήσουμε καταλήλως τις ε, αρμόδιες εθνικές αρχές και το προσωπικό τους όσον αφορά την προστασία των άγριων ειδών και την καταπολέμηση του σχετικού εγκλήματος, αλλά και σε αυτό το τομέα και στους άλλους τομείς αντιμετωπίζουμε και το φαινόμενο της διαφθοράς, ένα ζήτημα πολύ σοβαρό το οποίο καθιστά μη αποτελεσματική τη μάχη κατά της εγκληματικότητας εις βάρος των άγρων ειδών, ακριβώς επειδή εξαιτία των υψηλών φαινομένων διαφθοράς πολλές φορές καταφέρνουν οι εγκληματικές αυτές ομάδες να παρακάμψουν ή και να διαφθείρουν πολλές φορές τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει με την υφιστάμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε υποστήριξη προς τις αρχές των χωρών προέλευσης. Σαφώς αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει, αλλά μην ξεχνάμε ότι πολύ συχνά ανάλογα προβλήματα έχουμε και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε εσείς στην, στον Ανατολικό Αυτοδρόμο, διάβλο παράνομης διακίνησης άγρων ειδών που πολλές φορές τον παραβλέπουμε γιατί επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην ε, μεσογειακή οδό, δηλαδή ε, στον διάβλο εκείνο που ε, διακινούνται κυρίως εξωτικά ζώα από την Αφρική. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε παράνομη διακίνηση ειδών και από τη Ρασία και από την Ανατολική Ασία. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά περνάνε από αυτό τον Ανατολικό διάδρομο και πολλές φορές ακόμα και τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται σε αυτό τον ανατολικό διάβλο, σε αυτό τον ανατολικό διάδρομο δεν έχουν ε, τις απαραίτητες ε, αρχές ή τους απαραίτητους σπόρους προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα εγκληματικότητος. Και δύο ακόμα πράγματα θα θέλω να πω. Δεν έχουμε εθνικά σχέδια δράσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε σύντομα ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την εγκληματικότητα εις βάρος των αγρίων ειδών, αλλά δυστυχώς σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχο εθνικό σχέδιο δράσης. Απουσία λοιπόν τέτοιων εθνικών σχεδίων δράσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ευοδοθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης. Άρα να υιοθετήσουν τέτοια σχέδια και τα κρατημέλη και τελευταίο μου τώρα σχόλιο θα πρέπει η μάχη κατά της εγκληματικότητα, εις βάρος των άγρων ειδών να συνδεθεί με τους στόχους που έχουμε θέσει όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη. Ορισμένοι από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν την καταπολέμηση της λαθροθυρίας και την, παράνομη διακίνηση, την παράνομης διακίνησης άγρων φυτών και ζώων. Πρέπει λοιπόν να υποφεληθούμε τις ευκαιρίε που μας δίνεται αυτή τη στιγμή προκειμένου να αναρμονίσουμε τη δική μας τη δράση με τη δράση των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια της καταπολέμησης τη εγκληματικότητα ει βάρο των αγρίων ειδών. Για άλλη μια φορά σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και ελπίζω ότι σε μερικά χρόνια θα είμαστε σε θέση να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές επιτροπές, πάρα πολλά σχέδια δράσης. Το ζήτημα δεν είναι η θεωρία, αλλά η πράξη. Πώς θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε δηλαδή το σχέδιο αυτό δράσης. Ελπίζω λοιπόν ότι με τη βοήθεια των κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ένα αποτελεσματικό τέτοιο σχέδιο δράσης, το οποίο πραγματικά θα συμβάλλει στην πάταξη της εγκληματικότητας κατά των άγρων ειδών. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γνανό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 8 με 20 εκατομμύρια ευρώ περιέρχονται στα χέρια εγκληματικών ομάδων που ειδικεύεται στην ε, παράνομη διακίνηση άγρων ειδών και συνδέονται πάρα πολύ βέβαια οι ομάδες αυτές με τις παράνομες ομάδες διακίνησης ναρκωτικών, ανθρώπων κτλ. Απέναντι στα φαινόμενα αυτά δεν υπάρχει πανάκια, μία και μοναδική λύση. Νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να πλαισιώσουμε νομοθετικά με τον καλύτερο δυνατό αυτό τρόπο το πρόβλημα αυτό και να πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα εγκληματικότητα. Το καλύτερο είναι να μπορούμε ήδη στις χώρες προέλευσης, όπως στις χώρες της Αφρικής, να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του λαθρεμπορίου αγρίων ειδών. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές οι ομάδες αυτές εποφελούνται της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων αναπτυσσόμενων αφρικανικών χωρών. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να επιβληθεί καταλήλως η ε, δασοκομική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά συγκεκριμένες ζώνες προστασίας. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τις πιο ευαίσθητες γεωγραφικές ζώνες. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προστατεύσουμε συγκεκριμένα ίδια αν δεν θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του παράγωγου δικαίου έχει πιο δεσμευτικές διατάξεις σε σχέση με αυτές που προβλέπονται σε φυστάμενες διεθνείς συμφωνίες. Εμείς θεωρώ παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να ασκούμε πίεση προκειμένου όλες οι υπόλοιπες χώρες, οι τρίτες χώρες δηλαδή, να μπορούν να εφαρμόζουν ανάλογες με την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσίες οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται και στην πράξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πότς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Αναφέρατε ότι συνεργαστήκατε με πέντε χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η επιβολή του νόμου πραγματοποιείται από τα κράτη-μέλη. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω σε τι βαθμό ζητήσατε τις εμπειρίες από τη δική μου χώρα, την Σεχία, διότι έχουμε αρκετή επιτυχία όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Βλέπουμε ε, κατασχέσεις ε, ζώων. Δεν ξέρω λοιπόν γιατί χρησιμοποίησατε παραδείγματα μόνο από πέντε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μία ερώτηση στην οποία αναφέρθηκε και ο συνάδελφος. Θα προσπαθήσω να την διατυπώσω με ακρίβεια. Το νόμιμο εμπόριο εμποδίζει ή στηρίζει ε, το έγκλημα ε, εις βάρος των άγριων ειδών θα βοηθήσει την κατάσταση το να δημιουργήσουμε μια νόμιμη αγορά ή θα την επιδεινώσει. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι ευρωβουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Όχι. Τότε να ξαναδώσουμε το λόγο ε, στους συντάκτες της μελέτης. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις ε, τέθηκαν. και θα σχολιάσω και τις παρεμβάσει που έγιναν όπως και ο συνάδελφός μου άλλωστε. Ε, όσον αφορά το γιατί εξετάσαμε ει βάθο μόνο πέντε χώρε, επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Δεν εξετάσαμε την κατάσταση μόνο σε αυτές τις πέντε χώρε, εξετάσαμε και τις εκθέσεις site που καλύπτουν 25 κράτη-μέλη καθώ. και μελέτες από 25 χώρες. Ε, απλά εξετάσαν περισσότερο εις βάθος πέντε κράτη. Αυτό έχει να κάνει με το χρόνο και τον προπολογισμό που είχαμε στη διάθεσή μας. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε την κατάσταση σε διάφορα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, επειδή οι εμπειρογνώμονες ε, θεώρησαν ότι είναι κόμβοι ε, ή ότι είχαν ιδιαίτερη επιτυχία στην επιβολή του νόμου. Αλλά ναι, φυσικά θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει άλλες χώρες. Ε, πάντα πρέπει να διαλέξει κανείς. Νομίζω όμως ότι επιλέξαμε κράτη-μέλη αντιπροσωπευτικά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκαν και κάποιες άλλες ε, πτυχές το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος, για παράδειγμα. Ε, φιλολογία που εξετάσαμε μας δείχνει ότι ε, σε διάφορες μελέτες ε, καταδεικνύεται η σχέση ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και το έγκλημα εις βάρος των άγριων ειδών. Άλλοι εμπειρογνώμονες όμως θεωρούν ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν αποτελεί πρόβλημα όσον αφορά τα κλίματα εις βάρος των άγριων ειδών, ε, όπως ε, στην Γερμανία και στις κάτω χώρες. Ε, μπορεί λοιπόν αυτό να ισχύει σε κάποιε χώρε και μάλιστα σε κάποια κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτομάτω όμω ότι υπάρχει σχέση σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τα σχέδια δράση και τα ε, το αν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τέτοια. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα αυτό και να υπάρχουν σχέδια δράσης ε, από τα κράτη-μέλη που έχουν σχέδια δράσης ε, εξετάσαμε τις επιπτώσεις. Πάντως για κάποια κράτη-μέλη ήταν ε, ε, θεωρήθηκε σκόπιμο το να μην έχουν κράτη-μέλη. Ε, λήφθη σχετική απόφαση κατόπιν σχετικής μελέτης. Σε περίπτωση λοιπόν που ένα κράτος μέλος δεν έχει κράτος μέλος, σημαντικό είναι να εξετάσουμε το γιατί δεν δίνει προτεραιότητα στο θέμα ή υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί καταπολέμησης του προβλήματος. Μία ακόμα παρατήρηση πρωτού να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, κυρώσεις, διότι ο συνάδελφός μου είπε ότι δεν φαίνεται να είμαστε υπέρ της εναρμόνισης των κυρώσεων ε, στο έγκλημα εις βάρος των άγριων ειδών και ήθελα να εξηγήσω το γιατί. Εξετάσαμε τις κυρώσεις που επιβάλλονται και διαπιστώσαμε ότι απέχουν πολύ από το μέγιστο που επιτρέπεται και αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, το οποίο σημαίνει ότι αν τα δικαστήρια θέλουν να επιβάλλουν πιο αυστηρές κυρώσεις μπορούν να το κάνουν αυτό και αν ε, είναι ε, δυνατό Εάν ε, το μέγιστο είναι υψηλότερο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιβάλλονται στην πράξη υψηλότερε κυρώσει. Γι' αυτό θέλαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην επιβολή του νόμου, αντί να θεσπίσουμε έναν κανόνα, ο οποίο όμω δεν θα αλλάξει τίποτα στην πράξη. Να προσθέσω κάτι. Ποιος είναι ο λόγος που όσον αφορά την εναρμόνιση των κυρώσεων ε, συστήνουμε αυτό να γίνει στο πλαίσιο της οδηγίας ε, για την ε, για, το, ε, για το περιβαλλοντικό έγκλημα. Το θέμα μας είναι η σχέση και με άλλα θέματα. Εάν λοιπόν θέλουμε εναρμόνιση, αυτό θα πρέπει να γίνει γενικά στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού εγκλήματος και όχι αποκλειστικά στο τομέα του εγκλήματος κατά της άγριας πανίδας, διότι αλλιώς θα έχουμε υπερβολικά πολλά διαφορετικά καθεστώτα τα οποία δεν ταιριάζουν μεταξύ τους όσον αφορά το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπόθηκε ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Δεν ε, έχει στόχο η μελέτη μας να αξιολογήσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο δεν είχε τη θέση ισχύ ακόμα κατά την ολοκλήρωση της μελέτης μας. Στην ε, σύσταση του 2007 Αναφερόμαστε όχι μόνο στις κυρώσεις αλλά και στην πρόληψη και την γενική προσέγγιση, κάτι που αποτελεί βήμα προόδου. Αναφέρονται επίσης τα χρονοδιαγράμματα και η παρακολούθηση, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι θα μπορούσε να έχει κανείς ένα σχέδιο δράσης με πάρα πολλές συγκεκριμένες δράσεις, ε, αλλά που να μην εφαρμόζεται στην πράξη με λοιπόν ή χωρίς εθνικά σχέδια δράσης. Ε, θέλουμε να γίνει κάτι στην πράξη. Τα εθνικά σχέδια δράσης μπορούν ε, να βοηθήσουν την κατάσταση, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς την ύπαρξη τέτοιων σχεδίων. Η παρακολούθηση όμως και τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ σημαντικά θέματα όσον αφορά την πρόσθετη νομοθεσία. Δεν λέμε ότι θα ήταν περιττή αλλά είπαμε για παράδειγμα ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι παραπονέθηκαν ότι είναι υπερβολικά πολύπλοκη η νομοθεσία στο θέμα της άγριας πανίδας. Ε, δεν είναι πάντα ε, εύκολο κατανόητη και επίσης όσον αφορά πιθανά παραθυράκια στο νόμο. Συχνά οι διακινητές ε, περνούν ζώα τα οποία ε, έχουν ε, θύματα λαθροθυρίας ε, ως ζώα εκτροφής. Το σημαντικό μας πρόβλημα είναι η υποβολή του νόμου. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και όχι στη δημιουργία νέας νομοθεσίας, όπου μπορεί και πάλι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της επιβολής του νόμου. Και νομίζω επίσης δεν απαντήθηκε το ερώτημα σχετικά με την σχέση ανάμεσα στο νόμιμο και το ε, παράνομο εμπόριο. Ε, εάν δηλαδή δώσουμε την δυνατότητα για νόμιμο εμπόριο, μήπως ε, εξαλειφθεί έτσι το παράνομο εμπόριο. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ευρύ ερώτημα, έχει να κάνει με τα διάφορα είδη και τις διάφορες χώρες, ε, διότι είναι και διαφορετικά τα κίνητρα. Κάποιοι ενδιαφέρονται για το κέρδος, άλλοι για τα σπάνια είδη. Νομίζω ότι με βάση τις συνεντεύξεις ε, που είχαμε μπορούμε να πούμε ότι γίνεται πιο δύσκολη η επιβολή του νόμου επειδή κάποια είδη μπορούν ε, να ε, εκτραφούν και να τα εμπορεύεται κανείς νόμιμα ενώ εάν έχουν πιαστεί από την ε, φύση, τότε είναι παράνομη η διακίνησή τους. Επίσης, ε, η εκτροφή άγριας πανίδας ε, και η εμπορία της μπορεί να αποτελεί πηγή εισοδήματος σε κάποιες χώρες προέλευσης, αλλά Εάν εξετάσουμε και άλλους ε, τομείς εγκλήματος, όπου καθίσατε παράνομο το εμπόριο κάποιων ειδών, αυτό δεν σημαίνει κιόλας ότι σταματάει. Το να γίνει το εμπόριο γενικά παράνομο δεν θα το σταματήσει παρότι μπορεί να διευκολύνει κάπως την επιβολή του, νόμου. Πάντως ε, είναι πολύ πλοκό ερώτημα και έχει να κάνει με το για ποια χώρα μιλάμε, για ποιο είδος κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Ο αντιπρόεδρος μας ε, ζήτησε πάλι το λόγο. Υπόσχομαι ότι δεν θα μακρηγορήσω. Απλά να πω ότι αναφέρατε ότι είναι πιο σημαντική η επιβολή του νόμου από τη δημιουργία νέας νομοθεσίας, αλλά μερικές φορές σχετίζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, την πατρίδα μου, έχουμε ε, αρκετά αυστηρούς κανόνες σχετικά με το περιβαλλοντικό έγκλημα που θα πρέπει να αποτελεί το γενικό μας πλαίσιο. Δεν είναι όμως απόλυτα σαφές πώς θα εφαρμόζεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αγρία πανίδα επικεντρώνονται στη, στην ζημιά στη φύση και στο περιβάλλον. Εάν λοιπόν ο εισαγγελέα ή ο δικαστής θεωρήσει ότι η διακίνηση άγριων ειδών εμπίπτει στο περιβαλλοντικό έγκλημα, μπορεί αυτό να αρκεί, αλλά στην πράξη αυτό δεν γίνεται. Θα μπορούσαμε λοιπόν ενδεχομένως να ζητήσουμε καλύτερη επιβολή, αλλά μια διευκρίνηση εντός της νομοθεσίας που να λέει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρές κυρώσεις και στο εμπόριο άγριων ειδών, αυτό αποτελεί πτυχή της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε. Όπως προανέφερα, δεν είμαστε κατά της υιοθέτησης νομοθεσίας. Ε, είναι να θέμα ε, του να ε, βάλουμε περισσότερο βάρος πάνω σε αυτό και θα απαιτηθεί ε, διευκρίνηση για αυτό. Πάρα πολλοί παράγοντες φυσικά σκέφτονται, να υπά... σκέφτονται ότι η νομοθεσία είναι πολύ πολύπλοκη και θα απαιτηθεί κάποια διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε τους δύο ειδικούς για την παρουσίασή τους και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. το οποίο το οποίο είχαμε χθες κανονικά αλλά το μεταφέραμε για σήμερα αφορά την μεταφορά αποβλήτων και θα ακούσουμε αρχικά την Κομισιόν, οπότε νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της Κομισιόν και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στη συζήτηση με τα, ε, μέλη. Ε, το λόγο λοιπόν αρχικά έχει η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που και πάλι επαναφέρατε το συγκεκριμένο ζήτημα στην ημερήθησια διάταξη και υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο θα ήθελα ε, να αναφέρω είναι ε, ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το πόσο καλή είναι η Επιτροπή σας για τη διαχείριση του χρόνου και γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστώ που επαναφέρατε το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή αυτού, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Αρχικά τη μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε και στη συνέχεια αναφέρω μερικά από τα βασικά ζητήματα όσον αφορά τη μεθοδολογία. Αυτή είναι η τέταρτη αναφορά σχετικά ε, με τις μεταφορές, ε, μεταφορές αποβλήτων από το 2010 μέχρι και το 2012. Η αναφορά συνοδεύεται από έγγραφα. Η αναφορά λοιπόν βασίζεται σε δύο αναφορές ε, τις οποίες τα κράτη-μέλη πρέπει να καταθέτουν κάθε χρόνο. Το πρώτο είναι ένα, μία αντίγραφ, ένα αντίγραφο σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά εγγράφων και το επόμενο αφορά μια υποβολή που γίνεται στην Κομισιόν. Και παρόλο που η στατιστική αναφορά που αναφέρθηκε υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και αυτό οφείλεται σε δύο γεγονότα. Αφενός η αναφορά, οι αναφορές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία εργαζόμαστε. Η αναφορά λοιπόν της Κομισιόν δεν μας δίνει μια πλήρη εικόνα Όσον αφορά τα δεδομένα, παρόλα αυτά έχουμε δεδομένα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά. Τα δεδομένα λοιπόν τα οποία παραδόθηκαν από την πλευρά των κρατών μελών είναι ότι θα πρέπει να είναι τα ίδια. Η Eurostat λοιπόν αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό με τα κράτη-μέλη και κάνει προσπάθειες για να έχει τα δεδομένα μέχρι την επόμενη αναφορά. Σε αυτό το πλαίσιο η αναφορά της Κομισιόν περιλαμβάνει δεδομένα για την διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων δεν αναφέρεται στη μεταφορά δεδομένα μη επικίνδυνων δεδομένων ε, αποβλήτων. Δεν υπάρχει υποχρέωση από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνεται αναφορά αυτού και η μεταφορά σε μη κράτη-μέλη του ΟΑΣΑ απαγορεύεται. Όμως η αναφορά δίνει δεδομένο για την παράνομη μεταφορά και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη. Ποια είναι τα βασικά αποτελέσματα. Υπάρχουν τέσσερα δεδομένα. Πρώτον, η αναφορά δείχνει ότι από το 2000 μέχρι το 2012 τα απόβλητα έχουν αυξηθεί κατά 26%, 26 το 2009. Υπήρξε μία μείωση, ελαφρά μείωση, ίσως λόγω της οικονομικής κρίσης. Η μεταχείριση τώρα από το 2010 μέχρι το 2011 το 90% όλων των ε, επικίνδυνων αποβλήτων ε, βρισκόταν υπό υπεξεργασία στην ίδια χώρα από όπου προέρχονταν. Και παρόλο που τα περισσότερα απόβλητα υπόκειται επεξέργαση εντός της χώρας, η κατάσταση αυξάνεται συνεχώς και διπλασιάστηκε κατά την περίοδο 2001 μέχρι το 2009 όμως έχουν μειωθεί ελαφρά κατά την περίοδο 10-12 ίσως λόγω της κρίσης από περιβαλλοντικής άποψης η μεταφορά αυτών ε, ίσως δεν είναι κάτι κακό. Κάποια κράτη-μέλη έχουν καλύτερες εγκαταστάσεις ε, για την επεξεργασία τέτοιων αποβλήτων, ενώ αλλά δεν έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις και πολύ συχνά η πλησιέστερη ε, εγκατάσταση ίσως να βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλη το 95% των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων έλαβε χώρα μεταξύ των κρατών μελών και αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει μια αποτελεσματικότητα στο θέμα και δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη. Επιπρόσθετα γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έλαβε απόβλητα από τρίτες χώρες και η ποσότητα αυτών κατά την περίοδο αυτή ξεπέρασε το ποσό αυτών που εξήχθησαν κατά πέντε φορές. Όσον αφορά τις παράνομες μεταφορές, εδώ υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Η νομοθεσία που έχουμε απαγορεύει κάποιες μεταφορές προς αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες εκτός. από τα ε, κράτη-μέλη το 2014 και ανέστρεψε το βάρος της αποδείξης για, τα, για τις αποστολές ηλεκτρικών αποβλήτων μια σωστή εφαρμογή, αυτή, μια σωστή εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα έχει θετικά αποτελέσματα πιστεύουμε και για τα οχήματα τα οποία αποσύρονται οι οδηγίες που έχουν υιοθετηθεί για την εφαρμογή αυτών από το Σεπτέμβριο του 2011 δεν είναι δεσμευτικά, όμως η οδηγία που υιοθετήθηκε θεωρούμε ότι θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να περιορίσουν τον αριθμό των παράνομων μεταφορών αποσυρμένων αυτοκινήτων. Όμως η Κομισιόν αυτή τη στιγμή κάνει μια ε, πρωτοβουλία ε, ε e- πάνω σε αυτό το θέμα. Αν λοιπόν αξιολογήσουμε την εφαρμογή αυτών των μέτρων ε, για το, dump, dumping, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας λοιπόν αναμένονται κάποια στιγμή ε, μέσα στη φετινή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, είμαι διαθέσιμος για ερωτήματα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χάουσλινγκ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ καταρχάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, σημαντική και καλή αυτή έκθεση. Κάποια από τα στοιχεία αυτά είναι τρομακτικά. 150 κιλά επικίνδυνων αποβλήτων ανα πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε και ακόμα πιο τρομακτικό βρίσκω ε, την αύξηση των παράνομων εξαγωγών. Ε, σίγουρα πρέπει να ενεργήσουμε πολύ γρήγορα. Και όπως είπατε είναι πολύ πιθανότητα πραγματικά στοιχεία να είναι ακόμα υψηλότερα. πώς έχουν ε, τα πράγματα όσον αφορά τις προτεραιότητές μας, δηλαδή την ε, μείωση των αποβλήτων. Δεν είναι αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να συμπεριλάβουμε και στην κυκλική οικονομία. Να έχουμε δηλαδή ένα στόχο μείωσης των αποβλήτων. και τι δυνατότητες ανακύκλωσης ε, υπάρχουν των επικίνδυνων αυτών ε, αποβλήτων. Ε, τι το θέμα εάν η διάθεση των απορριμμάτων αυτών γίνεται με στον τρόπο. Και επίσης χρειαζόμαστε μια υποχρεωτική βάση δεδομένων και υποχρεωτική ανταλλαγή δεδομένων ώστε να έχουμε δεδομένα για, ως βάση για μελλοντικές εκθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να κάνω και εγώ ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη μελέτη σας αναφέρεται τα μη κατηγοριοποιημένα απόβλητα, μη ταξινομημένα απόβλητα, μικρό το ποσοστό αυτών, αλλά φοβόμαστε ότι μπορεί να περιέχουν κάποια επικίνδυνα απόβλητα. Τι εννοείται με αυτό το non-classified. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι. Επομένως, έχετε το λόγο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω καταρχάς στο δικό σας το ερώτημα. Αυτά τα μη ταξινομημένα, μη κατηγοριοποιημένα απόβλητα ουσιαστικά δεν αντιστοιχούν σε επικίνδυνα απόβλητα. Αυτό που συμβαίνει στην ουσία είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ονοματολογία για τα απόβλητα αυτά όσον αφορά τον κανονισμό για την διάθεση αποβλήτων, αλλά καταγράφονται από τα κράτη-μέλη, απλώς δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις υφιστάμενες κατηγορίες. Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την μικρή αυτή κατηγορία, non-classified. Τώρα, όσον αφορά τα αυξημένα ποσά επικίνδυνα αποβλήτων, Όντως, έχουμε αυξητική τάση. Εν μέρει αυτό οφείλεται και στη δική μας νομοθεσία που γίνεται όλο και πιο αυστηρή. Όσον αφορά δηλαδή την ταξινόμηση των αποβλήτων και τι χαρακτηρίζουμε επικίνδυνο και τι όχι. Και επίσης γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι όσον αφορά την επεξεργασία και τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων. Θεωρώ λοιπόν ότι τα όσα κάνουμε αυτή τη στιγμή μας επιτρέπουν να δεσμεύουμε πολύ περισσότερα επικίνδυνα απόβλητα και ότι δεν παράγουμε τελικά στην ουσία περισσότερα επικίνδυνα απόβλητα από ό,τι στο παρελθόν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο. Πρέπει να ασχοληθούμε και να περιορίσουμε τον αριθμό αυτών των επικίνδυνων αποβλήτων και στην, στον κανονισμό που παρουσιάσαμε τον Δεκέμβριο και στην έκθεση που περιμένουμε από τη δική σας Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και κάποιες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, απαιτήσει μάλλον προς τα κράτη-μέλη, να έχουν προγράμματα πολύ πιο αυστηρά και πολύ πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόληψη των αποβλήτων αυτών, γενικότερα των αποβλήτων και βέβαια σε αυτά περιλαμβάνονται και τα επικίνδυνα απόβλητα. Και εφόσον τα επικίνδυνα απόβλητα απαιτούν ειδική ξεχωριστή επεξεργασία, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με πολύ πιο αυστηρές νομοθεσίες και για την επεξεργασία. Επομένω, ένα κίνητρο παραπάνω για να μειώσουν την παραγωγή τέτοιων επικίνδυνων αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι και στα πλαίσια της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων την οποία προτείναμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή των επικίνδυνων αποβλήτων. Αν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τέτοιο σύστημα, τότε θα έχουμε και πολύ πιο ακριβείς πληροφορίες και κατά συνέπεια θα έχουμε πολύ πιο αξιόπιστες πληροφορίες, τις οποίες θα μπορέσουμε να κοινοποιήσουμε και προς Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό με τη σειρά του θα αποτελέσει κίνητρο για να έχουν πιο αυστηρή νομοθεσία και μειωμένη παραγωγή τέτοιων αποβλήτων κράτη-μέλη. Καλύτερη διασύνδεση επίσης πρέπει να έχουμε και όσον αφορά τα συστήματα μεταφοράς τέτοιων αποβλήτων. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια, ένα αρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών που νομίζω θα μας επιτρέψει να καταγράφουμε καλύτερα οποιαδήποτε μεταφορά αποβλήτων και επικίνδυνα αποβλήτων μεταξύ των κρατών μελών. Θα έχουμε δηλαδή μια σφαιρική εικόνα που θα μας επιτρέπει να συμπληρώνουμε όλα αυτά τα κενά πληροφοριών τα οποία εντοπίζουμε επί του παρόντος. Πολλές φορές ε, τα δεδομένα τα οποία μας έρχονται από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος ή από τα, τη Eurostat παρουσιάζουν κάποια κενά. Θεωρώ πάντω ότι με τι υφιστάμενε προτάσει και με τι μελλοντικέ νομοθετικέ προτάσει στου επόμενου 12 μήνε θα είμαστε σε θέση πλέον να έχουμε μέσα τα οποία θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θίξατε. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ χρήσιμη αυτή παρουσίασή της. Νομίζω ότι μπορούμε στο σημείο αυτό να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 23 και 24 Απριλίου, Μαΐου διορθώνει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Λύε τη σημερινή συνεδρία. Σας ευχαριστώ.